και, το, και την Επιτροπή μετά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 11 Φεβρουαρίου του 2015 σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση φασανιστήριων από την CIA. Θέλω να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου παράδοση. Σήμερα καλή παράδοση. Ο κύριος Κέντες έχει το λόγο. Thank you very much, uh, Mr. President. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Ευρωβουλευτέ, όπω γνωρίζετε, η ΕΠΑ είναι ένα σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Γνωρίζετε όλοι επίση ότι υπήρξαν διάφορες ανησυχίε και διαφορές στο παρελθόν σε σχέση με την αντιτρομοκρατική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιες πτυχές αυτές. Έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα πολλές, εδώ και πολλά χρόνια για σύνορα, για μεταγωγές, ε, ε, σε σχέση με τις διεθνείς προδιαγραφές και στάνταρ. Έτσι μπορέσαμε να θίξουμε διάφορα ζητήματα και σοβαρές ανησυχίες που έχουμε για το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τώρα είμαστε στο ΕΝΕΤΗ 2016 και ότι ο πρόεδρος Ομπάμα επισήμως σταμάτησε το πρόγραμμα της CIA λίγες μέρες μετά την ανάληψη καθηκόντων του που ήταν πολύ σημαντική απόφαση, κρίσιμη απόφαση. Μάλιστα, με δική του, δικό του διάταγμα απογόρευσε οποιοδήποτε είδος βασανιστήριων, καθώς και εκείνες τις τεχνικές που ονομάζονται ε, εντατικές τεχνικές ε, ανακρίσεων. Πιστεύουμε ότι τα βασανιστήρια είναι κατά των αξιών μας και δεν εξυπηρετούν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Το Συμβούλιο επανειλημμένα είπε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να γίνεται με, σε πλήρη σεβασμό του διεθνού, της διεθνούς νομοθεσίας, της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί προσφύγων. Αυτό ισχύει τότε και ισχύει και σήμερα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ιδρυμοκρατία μόνο αν μείνουμε πιστοί στι βασικέ μα ε, αξίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κάθε μορφή βασανιστηρίου και κάθε άλλη κακή μεταχείριση και οποιοδήποτε συνθήκε και εργάζεται κατά της πρόληψη και τη εκρίζωση του στην Ένωση αλλά και διεθνώ. Το πρόγραμμα που αναφέρθη σε, αυτό το, σε αυτή την ερώτηση έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια και ο πρόεδρος Ομπάμα έχει προσεγγίσει την αντιτρομοκρατική ε, πολιτική της, ε, τον ΗΠΑ σε αυτήν της Ένωσης. Είχε απαγορέψει και αυτές ε, τις φημιζόμενες εντατικές τεχνικές ανακρίσεων και αυτές απαγορεύθηκαν. Ορίζεται ότι η εθνική ασφάλεια βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρης ευθύνη κάθε κράτους μέλους. Αυτό σημαίνει ότι οι μυστικές υπηρεσίες κάθε κράτους είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της και γι' αυτό καταλαβαίνω κάποιες από τις ανησυχίες σας ότι το Συμβούλιο δεν έχει δώσει συνέχεια στις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο δικό σας ψήφισμα για τον απλό λόγο ότι το Συμβούλιο δεν έχει τις αρμοδιότητες να κάνει κάτι τέτοιο σύμφωνα με την συνθήκη της Ένωσης. Είναι ικανοποιητική αυτή η κατάσταση η απάντηση είναι πως όχι. Εγώ προσωπικά ως Ευρωπαίος ντρέπομαι που αυτές οι πρακτικές στο παρελθόν έγιναν, ε, έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος και θέλω να εκφράσω εξ ονόματος του Συμβουλίου την ίδια αυτή αίσθηση ντροπή. Όμως εμείς πρέπει να τηρήσουμε τις συνθήκες. Αλλά δεν είναι αυτό το τέλος. Είμαι βέβαιο ότι και η επίτροπο θα μπει σε κάποιες πτυχές που αφορούν τι δικέ αρμοδιότητες. Δεν σημαίνει αυτό πως οι δραστηριότητε μεμονωμένων κατών μελών που συμμετέχουν σε δραστηριότητε ή που περνούν χωρί έλεγχο. Τα κράτη της Ένωσης οφείλουν βάσει την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και με βάση το θεμελιώδη χάρτη ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ένωσης <clears throat> να ε, δίνουν εξηγήσει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξετάζει την υπόθεση αυτή ε, για τις παράνομες μεταγωγές δε σε μία τουλάχιστον απόφασή του, σε μία τουλάχιστον τιμιγορία του καταδίκασε αυτές τις πρακτικές σε ευρωπαϊκές χώρες και το Συμβούλιο θέλει να υπογραμμίσει την σημασία αυτής της σημαντικής νομολογίας ε, η απόφαση και η κρίση θα πρέπει να ε, ε, ε επαφείται στο, ε, στις αποφάσεις του δικαστηρίου και μόνο. Αυτά που συνέβησαν με τις μεταγωγές μπορεί να, ε, να μην συμβούν, εύχομαι να μην συμβούν ποτέ ξανά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και τώρα Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Άλμπρεχτ. Παρακαλώ, έχετε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ο σεβασμός ε, των θεμελιωδών ε, αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια καθοριστική αξία για μας και κάθε φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταδικάσει αυτές τις κακομεταχειρήσεις, τα βασανιστήρια, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλου είδους απάνθρωπη μεταχείριση, καθώς και τις παράνομες κρατήσεις ε, θεωρώντας βεβαίως ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να εξαιρεθούν αυτές οι αξιόπινες πράξεις από την τιμωρία και την καταδίκη. Θεωρούμε ότι αυτού του είδους οι παράνομες κρατήσεις, οι μυστικές κρατήσεις θα πρέπει να απαγορεύονται και σε κάθε περίπτωση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει η πολιτική μας να βασίζεται στο κράτος δικαίου. Γι' αυτό και ζητούμε να υπάρξουν εντελεχείς έρευνες καθώς και η κάθε είδους συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και των απελάσεων που έλαβαν χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν όλα τα νέα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν και να υπάρξουν οι απαραίτητες έρευνες. Η έκθεση της Επιτροπής ε, της ε, Αμερικανικής Γερουσίας οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφοριών οι οποίες συνεργάστηκαν και έπαιξαν ρόλο σε αυτές τις παράνομες κρατήσεις. Πολλές φορές αυτό έγινε με την χρήση ε, παράνομων μέσων διαφθοράς και η έκθεση της Γερουσίας και των υπηρεσιών πληροφοριών απέδειξαν ότι χρησιμοποιήθηκαν ε, διάφορες ε, τεχνικές ε, ανάκρισης μεταξύ των οποίων και βίες. Η μαζική παρακολούθηση, το μαζικό πρόγραμμα παρακολούθησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε σαν στόχο πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει επίσης αποκαλυφθεί και γνωρίζουμε σήμερα ότι όσον αφορά την συνεργασία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ε, πληροφοριών υπήρξε σε πολλά επίπεδα συνεργασία. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπήρχε μυστική παρουσία σε ευρωπαϊκές χώρες ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει νέα στοιχεία για παράνομες κρατήσεις, για απελάσεις θα πρέπει να εξηχνιαστούν, να ερευνηθούν και να προσφύγουν όταν υπάρχει αντικείμενο στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Θεωρούμε ότι τα προγράμματα DCA, ο απόρριτος χαρακτήρας αυτών των υποθέσεων καθώς και η ατιμορρησία και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει παραβίαση μεταξύ της δικασικής συνεργασίας, μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανικών αρχών και σε κάθε περίπτωση παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης της υπερατλαντικής κάτι που διαπιστώνουμε ότι υποχρεώνει σήμερα τα ευρωπαϊκά κράτη να αντιδράσουν. Εμείς βεβαίως και στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες έρευνας και εξυχνίασης αυτών των υποθέσεων με τη χρήση όλων των απαραίτητων μέσων υπηρεσιών πληροφοριών έτσι ώστε να αποσαφινιστεί εάν υπήρξαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να καθοριστούν οι ρόλοι των υπηρεσιών πληροφοριών και των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων. Προτείνουμε να υπάρξουν συμφωνίες ε, για τις διασυνοριακές ε, αυτές επιχειρήσεις η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να θεωρηθεί ότι ξεπερνάει την νομοθεσία και το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Ε, ήθελα να σας ζητήσω να μιλάτε λίγο πιο αργά για να προλάβουν οι διερμηνείς αυτά που λέτε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούροβα, καλωσορίζω τι συνεχεί προσπάθειε του Κοινοβουλίου να παρακολουθήσουν το θέμα αυτό. Οι πρακτικέ που αναφέρονται στην έκθεση τη Γερουσία για, ε, για το πρόγραμμα κράτηση και ανάκριση τη CIA αποτελούν σοβαρά παραδείγματα παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όμως τονίζω ότι τα θέματα εθνικής ασφάλειας είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Η, Επιτροπή, η συνθήκη δίνει στην Επιτροπή αρμοδιότητες να ερευνά τη δράση των εθνικών υπηρεσιών ασφάλειας και την κατασκοπίας. Επιπλέον, ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων εφαρμόζεται μόνο όταν τα κράτη υλοποιούν νομοθεσία της Ένωσης. Τα γεγονότα που αναφέρονται είναι θέματα που βρίσκονται εκτός Ένωσης. Παρά τα αυτά ωστόσο η Επιτροπή υπογράμμιζε έκτοτε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει, τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν σε έρευνα για την εξέταση των γεγονότων και να επιτρέψουν στα θύματα να ζητήσουν αποζημίωση. Αυτό είναι μια θετική υποχρέωση που προκύπτει από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το υπενθύμησε και το ΕΔΑΔΑ. Σε ό,τι αφορά την δικαστική συνεργασία, την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε σχετική διάταξη στη σχετική διάταξη μεταξύ ΙΠΑ και Ένωσης. Υπήρχαν δύο συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την έκδοση και την αμοιβαία νομική συνδρομή, αλλά αυτές τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου του 2010 που ενοποιούν το νομικό θεσμικό πλαίσιο τη συνεργασία σε ποινικά ζητήματα με τη ΣΥΠΑ. Ομοίω την περίοδο των ε, γεγονότων δεν υπήρχαν ε, ε, ρυθμίσεις της Ένωσης για τον προσδιορισμό ατόμων ως προσφύγων, ούτε διαδικασίες χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα στην Ένωση. Η οδηγία 2004 του 83 και 2004-85 τέθηκαν σε ισχύ και ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία μετά τα γεγονότα. Μέσα στα πλαίσια της ενωσιακής νομοθεσίας ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να σέβονται πάντα τα πρότυπα των θεμελών Την ε, και στην συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και οπουδήποτε αλλού, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να υλοποιούν την Ομοθεσία για την δημοκρατία με συμβατό τρόπο σε σχέση με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Για τις πολιτικές ομάδες το λόγο έχουν οι εκπρόσωποι για το ΕΛΚ. Η κυρία Μετσόλα. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορούμε να χάνουμε το ευρύτερο πλαίσιο και τους στόχους μας και τι θέλουμε να προστατεύσουμε. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να προστατεύσουμε. Αξίες, ελευθερίες, δικαιώματα που θεωρούμε ότι κάποιες φορές απειλούνται στην Ευρώπη. Εμείς αρνούμεθα την τρομοκρατία γιατί αρνούμεθα να παραχωρήσουμε, να αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μας. Αυτό είναι που μας κάνει Ευρωπαίους. Η χρήση βασανιστήριων αντιβαίνει ευθέως στις αξίες που περασπίζουμε. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ποτέ. Δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Τα βασανιστήρια δεν θα επιτρέψουν δεν μας επιτρέψουν ποτέ να αισθανόμαστε άνετοι. Η μάχη κατά της δημοκρατίας πρέπει να είναι αποτελεσματική, αλλά πρέπει να είναι ταυτόχρονα ισορροπημένη και να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αρχές μας στις δύσκολες στιγμές. Αντίθετα, σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να διπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας. Γι' αυτό ξεκίνησε η Εξεταστική Επιτροπή πέρυσι, ούτω ώστε να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος και να μην τα επαναλάβουμε. Τα βασανιστήρια δεν μπορεί να είναι το όπλο μας, δεν εκφράζει αρχές μας, ούτε αυτά που πιστεύουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών, η κυρία Φάγιον. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Ευρωκοινοβούλιο ζητούμε από τα κράτη-μέλη να λάβουν σοβαρά μέτρα. Η έκθεση της Γερουσίας ε, των είπα, αποκάλυπτε ότι η CIA ε, προέβησε βασανιστήρια και, και χρησιμοποίησε βίες μεθόδους ανακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευρωπαϊκών αξιών. Νέα στοιχεία προκύπτουν με την αντιπροσωπεία της ΛΥΜΠΕ επισκεφθήκαμε τη Ρουμανία πέρυσι, αλλά οι αρχές δεν μας επέτρεψαν να μπούμε στο κτίριο όπου κρατούνταν οι ε, κρατούμενη εκείνη την εποχή. Ε, και η Λιθουανία ε, ε, ε, συνέβαλε στην αποκάλυψη στοιχείων. Αυτό όμω, που ήταν καθοριστικό ήταν η εμπιστευτική έκθεση τη Αμερικανική Γερουσία, που όχι μόνο αποκάλυψε τη διάσταση των εγκλημάτων αλλά και το γεγονό ότι τα βασανιστήρια δεν είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση τη τρομοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα βασανιστήρια και πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί ω προ αυτό. Πρόκειται για συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων και ανθρωπιστικών δικαιωμάτων, την πιο σοβαρή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο ε, Πόλεμο. Οι δε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους. Είναι λυπηρό που οι η βιομηχανία ταινιών του Χόλιγου ήταν αυτή που είχε τα περισσότερα στοιχεία για αυτά τα βαστινιστήρια. Ακόμα και οι δικηγόροι των κρατουμένων δεν κατάφεραν να έχουν αυτά τα στοιχεία και οι διάφοροι άνθρωποι, ε, κρατούμενοι υπάρχουν ακόμα στον στο Γκουαντάναμο, φυλακισμένοι, χωρίς να έχουν ε, περάσει από, καν από δίκη. Οι έρευνε πρέπει να συνεχιστούν, να ξέρουμε πόσα κράτη συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία. Αυτές οι παραβιάσεις δεν θα εξαφανιστούν και κανένα ένα δεν είναι αρκετά μεγάλο ώστε να τα ε, κρύψουμε όλα αυτά από κάτω. Ε, πρέπει λοιπόν να ρίξουμε άπλο το φως σε αυτή την πολύ ντροπιαστική στιγμή της ιστορίας μας και να εξασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Θέλω να κάνω έκκληση σε όλους τους συνάδελφους ώστε να είμαστε ενωμένοι αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ που μείνατε εντός του χρόνου σας. Τώρα εξ ονόματος του ECR το λόγο έχει ο κύριος Ουγιασδόφσκι. Κυρίες και κύριοι, ένας πολιτισμένος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να κατακρίνει την τρομοκρατία, την αυθαίρετη κράτηση και άλλα έκτακτα μέτρα, αλλά εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται τώρα αυτό το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπε και ο Υπουργός, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, καταρχάς οι Ηνωμένε Πολιτείε σταμάτησαν το πρόγραμμα αυτό που μπορεί να γεννά επικρίσει, αμφιβολίες και μπορεί να έχει ανάγκη περαιτέρω έρευνα. Η κυρία Γιούροβα είπε ότι η Ένωση δεν είχε τότε νομικά εργαλεία στη διάθεσή της, ούτε υπήρχαν συμφωνίες ή άλλα νομικά κείμενα. Η Προεδρία θύμισε ότι το θέμα της εθνικής ασφάλειας αποτελεί η αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και εκεί πρέπει να γίνει δουλειά για να εξεταστούν τα γεγονότα. Τέλος, το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες, αλλά έχει το δικαίωμα να ερευνά κάτι τέτοιο βάσει των συνθήκων. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο εναντί ευρωπαϊκών οργάνων, όχι εναντί, εναντί κρατών μελών. Άρα πρέπει να έχουμε μια πιο ορθολογική προσέγγιση στην δράση μας. Βεβαίως, δεν μπορεί να διαφορούμε ενώπιον ε, της χρήσης μη πολιτισμένων μεθόδων όπως των βασανιστήριων. Αλλά στη συζήτηση αυτή δεν, γίνεται, δεν μιλάμε για τρομοκράτες. Ε, γιατί δεν μιλάμε για τρομοκράτες. Οι τρομοκράτες θέλουν να καταστρέψουν τον πολιτισμό μας. Προφανώ δεν μπορούμε να χτυπάμε τους τρομοκράτες καταχρώμενοι των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αλλά ούτε μπορούμε να ερμηνεύουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου, ούτω ώστε να παραλύει ο ελεύθερο κόσμο όταν αγωνίζεται να χτυπήσει την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιντεβέλ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ήμουν μέλος της Επιτροπής Έρευνας ε, για το πρόγραμμα μεταγωγών της CIA. Πριν από 10 χρόνια περίπου έγιναν όλα αυτά. Και θα έλεγε κανεί μετά από 10 χρόνια, μα γιατί το συζητάμε ακόμα αυτό το θέμα και επαναλαμβάνουμε τις ίδιες δηλώσεις. Και πρέπει να σας πω ότι ποτέ, ποτέ δεν θα σταματήσω να ασχολούμαι αυτό το θέμα μέχρι ό,τι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μπορούμε να μιλάμε για το αν ίσχυε το ίδιο νομικό πλαίσιο τότε ή αν είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Ε, πάντως εγώ έχω την αίσθηση ότι το Συμβούλιο και τα κρατημέλη κρύβονται πίσω από νομικίστικα επιχειρήματα. Γιατί, Υπουργέ Κούντερς, αν είναι αλήθεια ότι η εθνική ασφάλεια είναι απλά και καθαρά εθνικό ζήτημα, τότε γιατί τα, τα, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, και αν θυμάμαι καλά ήταν τον Οκτώβριο του 2001, συλλογικά αποφάσισαν να επιτρέψουν τις πτήσεις αυτές της CIA από τον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο. Συλλογικά το αποφάσισαν αυτό και τώρα κρύβονται πίσω από αυτό το επιχείρημα. Λέγοντας, όχι, όχι, είναι εθνικό θέμα. Ενώ πρόκειται για λογοδοσία και ευθύνη, ε, τώρα ξαφνικά είναι εθνικό το ζήτημα. Όχι, αν οι κυβερνήσει τότε είχαν το θάρρο να λάβουν αυτή την απόφαση συλλογικά, τότε θα έπρεπε και τώρα συλλογικά να είναι ε, υπόλογοι και υπεύθυνοι. Όχι να κρύβονται πίσω από αυτά τα επιχειρήματα και να λένε Έχουμε τώρα ένα, λέει, ε, πολύ στερεό δικαστικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο. Εγώ όμως είδα ότι τις εθνικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως χρώματος, έκαναν ό,τι μπορούσαν ώστε να εμποδίσουν τις δικαστικές έρευνες και τις διώξεις. Έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους ώστε να σταματήσουν αυτές τις διαδικασίες. Και εσείς αναφέρατε τη λέξη ντροπή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Είναι τρομερή ντροπή δέκα χρόνια μετά από την πρώτη έκθεση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλάμε για το ίδιο πράγμα και είναι σαν να... Σαν να μιλάμε σαν ένα τείχο. Κανεί δεν μας ακούει. Εμείς όμως θα επαναρχόμαστε διαρκώ μέχρι ότου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν επιτρέπεται η αδημορρησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό, Υπουργέ Κούντερ, αυτό είναι ντροπή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βερσιά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, εδώ και δέκα χρόνια εργαζόμαστε σαν κοινοβούλιο σε αυτές τις ε, υπόνοιες για παράνομες κρατήσεις και παράνομες δραστηριότητες της CIA. Και βεβαίως υπάρχουν αρχές και κυβερνήσεις που εμποδίζουν τις εργασίες μας. Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σοβαρές και αυτό έγινε, έχει αποδειχθεί και φυσικά ακόμα και η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το έχει δηλώσει. Δεν μπορούμε εδώ να κρυβόμαστε πίσω από τις ε, συμφωνίες και τις συμβάσεις. Τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν σε πραγματικές έρευνες. Θέλουμε να γνωρίσουμε την αλήθεια έτσι ώστε τα θύματα επιτέλους να μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να δικαιωθούν. Τίποτα δεν δικαιολογεί τα βασανιστήρια. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να εκφράσω την ε, ε, λύπη μου, διότι παρόλες τις δηλώσεις του Προέδρου Ομπάμα, συνεχίζει να λειτουργεί το κέντρο κράτησης του Κουαντάναμου και άνθρωποι να κρατούνται εκεί παράνομα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βερζιά. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό η μπλε κάρτα μπορεί να υποβληθεί από κάποιον που δεν είναι στον κατάλογο των ομιλητών. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Εύα Ζολή για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το Δεκέμβριο του 2014 η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε μια έκθεση η οποία επιβεβαιώνει την συνεργασία πολλών κρατών ομελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις ε, δραστηριότητες κάτι που αποδεικνύει ότι το 2001 2006 υπήρξαν ε, τέτοιες δραστηριότητες και βασανιστήρια στην επικράτεια πολλών ευρωπαϊκών κρατών. Η δράση λοιπόν των ευρωπαϊκών κρατών και των θεσμικών τους οργάνων κατά εκείνη την περίοδο ήταν απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την, ατιμορα... στην ατιμορρησία εν ώψη τέτοιων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να συνεχιστούν οι έρευνες και οι ανακρίσεις και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτές οι απαράδεκτες παραβιάσεις, πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συνεχιστούν. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταδικάσουμε αυτές τις ε, περιπτώσεις όπου συνεργάστηκαν σε τέτοιες υποθέσεις ε, ευρωπαϊκά κράτη. Οι ανακρίσεις, οι έρευνες θα πρέπει να συνεχιστούν και μέχρι να υπάρξει πλήρης αποκάλυψη της αλήθειας δεν θα πρέπει να σταματήσουν γιατί πρόκειται για την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για την τιμή της Ευρώπης. Ελπίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, να υποστηρίξετε αυτή τη διαδικασία μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζολή. Και τώρα, εξ του EFTT, ο κύριος Καράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, ας το πούμε ξεκάθαρα. Είναι πραγματικά ντροπή. Είναι ντροπή που ε, μετά από σχεδόν 15 χρόνια, ενώ εγκρίθηκε ψήφισμα από αυτό εδώ το κοινοβούλιο πριν από 1,5 χρόνο ξανά, δεν υπήρξε καμία στήριξη, δεν ξεκίνησε καμία έρευνα. Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να κρύβονται πίσω από το ε, ρυθμιστικό πλαίσιο ή πίσω από τα κρατικά απόρριτα στοιχεία. Ε, στη στιγμή που δεχόμαστε εντό ε, των κρατών μελών μα, γιατί έγινε στη Ρουμανία, στην Πολωνία, έγινε στη Λιθουανία, και αυτό έχει επικυρωθεί από την έκθεση της Αμερικανικής γερουσία Στη στιγμή που δεχόμαστε λοιπόν να, έρχονται, να γίνονται μάλλον ε, βασανιστήρια, να γίνονται από άνθρωπες ε, ανακρίσεις, αυτό μπορεί να συμβεί σε καθέναν από εμά. Ήρθε η στιγμή να υψώσουμε τη φωνή μας και να ζητήσουμε οι ένοχοι να πληρώσουν, γιατί προχωρώντας έτσι δεν θα φτάσουμε πουθενά. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, Παπαδάκης, εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων. αβίαστο είναι το συμπέρασμα από τις αποκαλύψεις για τα φρικτά βασανιστήρια της cia σε κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης στον Κουαντάναμο και στις Ηνωμένε πολιτείες. οι Ηνωμένε πολιτείες η ευρωπαϊκή ένωση και οι κυβερνήσεις της που ευθύνονται έμειναν και μένουν στο απειρόβλητο. οι επιτροπές που στήθηκαν ήταν κυριολεκτικά για να ξεπλύνουν τις ευθύνες των υπεριαλιστών. πάει πολύ να προβάλλεται την ευρωπαϊκή ένωση ως υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την ίδια στιγμή που καλείται σε ενίσχυση της λεγόμενης αντιτρομοκρατική συνεργασίας με τις Ηνωμένε Πολιτείε στο όνομα τη οποία πραγματοποιείται υπεριαλιστικούς πολέμους και βασανιστήρια κατασταλτικοί μηχανισμοί των ηνωμένων πολιτειών της ευρωπαϊκής ένωσης του νατο και υπηρεσίες όπως η cia ο ευρωστρατός η κέπα η europol η νέα συνοριοφυλακή ακτοφυλακή συνεργάζονται στενά για το χτύπημα του λαϊκού κινήματος την καταστολή προσφύγων και μεταναστών ανταγωνίζονται στην κρατική και βιομηχανική κατασκοπία για τα κέρδη των μονοπωλίων τους. οι ίδιοι χρηματοδότησαν την αποκρουστική δράση μηχανισμών όπως το ισλαμικό κράτος. οι λαοί μπορεί να αχρηστεύσουν τους αντιδραστικούς μηχανισμούς που υπερασπίζονται την καπιταλιστική βαρβαρότητα παίρνοντας οι ίδιοι την εξουσία και την ιδιοκτησία του πλούτου που παράγουν. Ε, ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ. Μακάλιστερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, τα βασανιστήρια δεν μπορεί να δικαιολογηθούν υπό καμία προϋπόθεση. Ούτε και αυτές οι πρακτικές ε, βίες ανακρίσεων όπως αναφέρθηκαν από τη Γερουσία. Οι ΙΠΑ παίζουν κρίσιμο ρόλο στην καταπολέμηση τη τρομοκρατίας στον κόσμο και εδώ στην Ευρώπη. Η συνεργασία μα θα πρέπει να συνεργαστεί ε, για το κοινό καλό των πολιτών στι δύο όχθε του Ατλαντικού με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Χρειαζόμαστε συνεχιζόμενο πολιτικό διάλογο με του εταίρου μα για την ασφάλεια και την αντιτρομοκρατική δράση καθώ και για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την τρομοκρατία. Σε καιρούς παγκόσμιας ε, αστάθειας ε, αυτή η ατλαντική σχέση είναι πολύ στρατηγική σημασία και φύσης. Έχοντας υπόψη την έκθεση της Γερουσίας ε, για τη χρήση βασανιστήριων από τη θέλω να υπογραμμίσω τη δήλωση της 15ης Ιουνίου 2009 για το κλείσιμο του Guantanamo Bay και για τη μελλοντική αντιτρομοκρατική συνεργασία. Κοινέ προσπάθειες για τη τρομοκρατία θα πρέπει να συμβαδίζουν με τη διεθνή νομοθεσία, ιδιαίτερα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως τα δικαιώματα σε ανθρώπινη μεταχείριση, δίκαια δίκη και έλλειψη βασανιστήριων. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξαίρεση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκόμες. Παρακαλώ. Τα, οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Αμπούζο κατά Πολωνίας ενώ υπάρχουν αντίστοιχες ε, εκκρεμείς υποθέσεις κατά της Λιτουανίας και της Λετωνίας. Μια σειρά δικαστικών αποφάσεων στην Βρετανία είναι υπέρ των θυμάτων ε, των βασανιστήριων. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσει είπαν ψέματα στο Κοινοβούλιο για να καλύψουν με θρασί τρόπο παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στην η συνεργασία τους πληρώθηκε με μεγάλα ποσά. Το είπε η έκθεση της Γερουσίας. Ακόμα χειρότερο, είναι το ότι δόθηκε ατιμωρησία από τα κράτη της Ένωσης στους υπεύθυνους των εγκλημάτων αυτών. Για παράδειγμα, στην Ιταλία χρησιμοποιήθηκε το απόρριτο του κράτους για να παρεμποδιστεί η δικαιοσύνη. Αποτέλεσμα, καταδικάστηκαν ε, χαμηλόβαθμοι αθώοι ε, υπάλληλοι, ενώ οι υψηλόβαθμοι παρέμειναν στο απειρόβλητο. Μία ε, πολίτης, ε, μία πολίτης υπάλληλος τη CIA δικάστηκε ε, ερήμην χωρίς να μπορεί να, υπο, να παρουσιάσει την άποψή της. Στην περίπτωση ενός ενός ε, πολι... στην περίπτωση αυτή ένας από τα θύματα ο Αμπού Ομάρ δήλωσε ότι ήταν, χρησιμοποιήθηκε ως εξυλαστήριο θύμα. Στην Πορτογαλία χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αυτό και έκλεισε για να αποφευθεί να παραπεμφθεί ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν που ήταν πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Πώς θα πείσουμε τους πολίτες μας ότι τα κράτη χτυπούν την τρομοκρατία όταν κάνουν αντίστοιχα εγκλήματα. Θα συνεχίσω να ζητώ μέχρι τέλους να δοθεί να αποδοθεί δικαιοσύνη στο θέμα αυτό. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας. Η κυρία Άντερσον, ένα λεπτό. Η Διεθνής Αμνηστία επιβεβαίωσε ότι το αεροδρόμιο Σάνων στην Ιρλανδία χρησιμοποιήθηκε από τη ΣΥΠΑ και τη, και CIA για πτήσεις έκτακτων παραδόσεων. Χρησιμοποιήθηκαν ε, τεχνικές ε, βασανιστήριων που σύμφωνα με το ΕΔΑΔ ε, κρίθηκε ότι οι 14 Ιρλανδοί υπέστησαν απάνθρωποι μεταχείριση αλλά όχι βασανιστήρια. Αυτό επέτρεψε στην κυβέρνηση Μπούς να χρησιμοποιήσει τις πέντε τεχνικές βασανιστήριων. Ωστόσο οι Βρετανοί είπαν ψέματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας δεν κλήθηκε για περαιτέρω εξηγήσεις. Οι 14 Ιρλανδοί υπέστησαν φρικτές ε, ανακρίσεις από τις οποίες ποτέ δεν ανέκαμψαν. Εκατοντάδες παρόμοιες έκανε η CIA. Υπήρξαν βασανιστήρια, υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας και αυτή η εγκληματική συμπεριφορά πρέπει να εκτεθεί και να αμφισβητηθεί ούτως ώστε να αποφύγουμε τουλάχιστον να χρησιμοποιούν τα βασανιστήρια άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτσο. Ο κύριος Μπάλτσο είναι Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντως, εδώ και δέκα χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με τις επιχειρήσεις αυτές της CIA καθώς και τις παράνομες μεταγωγές, παραδόσεις κρατουμένων από την Ευρώπη στις Ηνωμένε Πολιτείε. Σε όλα τα έγγραφα που διαθέτουμε υπάρχει η λέξη καταγγελίες. καταγγελίες ή κατηγορίες και κάθε φορά βλέπουμε ότι το απόρριτο χρησιμοποιείται για να μην προχωρήσουν οι έρευνες. Κάθε φορά επίσης δεν κατονομάζονται οι Ηνωμένε Πολιτείες. Μιλάμε πάντα για CIA. Η CIA όμως δεν είναι χώρα. Θα πρέπει πραγματικά η αλήθεια να αποδειχθεί και να υπάρξουν οι συνέπειες για όλους τους ενόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λέναρτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το σημείο αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω την ε, απέχθειά μου για όλες αυτές τις ε, πρακτικές, τις κακομεταχειρήσεις, μέθοδοι βασανιστήριων απεχθείς που πραγματικά ποτέ, ποτέ δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Είναι δραματικά αυτά που συνέβησαν και συμφωνώ απολύτως με τους ε, συναδέλφους που ζητούν να υπάρξει αλήθεια, φως και να προχωρήσουν οι ε, έρευνες. Κοιτάξτε τα απογοητευτικά αποτελέσματα των προσπαθειών μας τις δύο τελευταίες ε, χρονιές μετά δηλαδή την ίδρυση της Επιτροπής. Ας είμαστε ρεαλιστές. Θα πρέπει αυτή η υπόθεση να συνεχιστεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και όπου αλλού μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Ε, συμφωνώ εδώ με τους συναδέλφους ε, από την ομάδα των φιλελευθέρων. Εμείς δεν στείλαμε παρά μία αποστολή κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν μόνο 70 από τα 70 μέλη συγγνώμη, των φιλελευθέρων μόνο ε, ένας να συμμετέχει σε αυτήν την αποστολή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήδη εδώ και χρόνια μιλάμε για αυτό το θέμα. Η μυστικότητα που περιβάλλει αυτό το πρόγραμμα εξ αρχής πολύ μας καθυστέρησε στο να καταλάβουμε τι έγινε ακριβώς και μόνο πολύ αργά μπορέσαμε να δούμε ποιον βαράνε οι ευθύνε και ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα πάντα. Ε, πρέπει αυτό να το πούμε και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το τι γίνεται σεβόμενοι την αρχή της επικουρικότητας και εκεί όπου πρέπει και βεβαίως προσπαθώντας να ξεκαθαρίσουμε το πολιτικό τοπίο. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως ιδεολογική προπαγάνδα. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τον συνομιλητή μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και δεν θέλουμε μόνο να ξεκαθαρίσουμε και να, να, να ε, αποδώσουμε ευθύνε. Αυτό που μας κάνει να συνεχίζουμε είναι ότι δεν πρέπει τέτοια πράγματα να ξαναγίνουν στο μέλλον. Θεωρούμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η τήρησή τους θα πρέπει να επικρατεί όλων των καταχρήσεων ε, των κρατών. Είναι μια αποστολή που πρέπει να συνεχίσουμε σε ε, ε, σεβασμό του παρελθόντος που δεν έχει ακόμα τελείως φωτιστεί και στο όνομα ενός μέλλοντος που το θέλουμε να είναι καλύτερο και να σέβεται περισσότερο τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα δικαιώματα του ανθρώπου, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Πρέπει να υπάρχουν και στην εθνική και διεθνή πολιτική της Ένωσης. Η καταπολέμηση της δημοκρατίας σημαίνει να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια του ανθρώπου όλα υπάγονται στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει την, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και την ασφάλεια των πολιτών τους. Η συνεργασία, η συνεργασία μεταξύ των κρατών πρέπει να γίνεται βάση κοινών αξιών. Η υπερπολιτικοποίηση ωστόσο του θέματος αυτού για την παράνομη κράτηση και την εμπλοκή της CIA σε κάποιες ε, διαδικασίες σύλληψης και παράδοσης ε, από ευρωπαϊκά κράτη προς τη ΣΥΠΑ μπορεί να ε, δημιουργήσει προβλήματα. Είναι καθήκον μας να επιστρέψουμε στα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν τις έρευνές τους και να μην εμπλακούν σε νομικές, σε δίκες που έχουν ξεκινήσει σεβόμενη την αρχή της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να δείξει ότι πρέπει να έχουμε στέρεες αποδείξεις πριν αρχίσουμε να καταγγέλουμε τους ε, κάποιους. Ευχαριστώ. Τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία Catch Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταδικάζουμε τις πρακτικές των βασανιστήριων από τη CIA στον Κουαντάναμο και σε άλλα κολαστήρια. Το σύστημα των μυστικών κρατήσεων της CIA οδήγησε σε μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε φρικτά βασανιστήρια. Οι μυστικές κρατήσεις της CIA περιελάμβαναν απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, βασανιστήρια, απαγωγές και κρατήσεις χωρίς δίκη. η χρήση βασανιστήριων δεν επιτρέπεται και βέβαια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να νομιμοποιηθεί για κανένα λόγο ούτε βέβαια για τη δίθεν αποκάλυψη πληροφοριών για το χτύπημα της τρομοκρατίας. φυσικά η ατιμορρυσία σχετικά με τις τακτικές που ακολουθεί η cia επιτρέπει τη συνέχιση της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο η ευρωπαϊκή ένωση να καταδικάσει κάθε μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβε χώρα από τη cia καθώς και να φροντίσει να διεξάγει περαιτέρω έρευνες σχετικά με τα κράτη μέλη της τα οποία σύμφωνα με την έκθεση ήταν συνένοχα στο πρόγραμμα μυστικών υπηρεσιών και εκτάκτων παραδόσεων της cia. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Θυμηθείτε πρώτα πρώτα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι σύμμαχος. Παρόλο που ο πρόεδρος της πρόσφατα παρενέβη στα εσωτερικά της Βρετανία. Η CIA δεν είναι υπό τον έλεγχο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευτυχώς ούτε και η MI5 υπηρεσίες ε, ασφαλείας και λιγατοσκοπίας θα πρέπει να ανακρίνουν με όσο πιο ανθρωπινό τρόπο γίνεται. Δεν πρέπει ωστόσο ο κόσμος να παρεμποδίζεται από πολιτικές αρχές σε βαθμό που να οδηγεί σε κίνδυνο. Το δικαίωμα στην ελευθερία δεν πρέπει να διακυβεύεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς δεν μπορούμε τους τρομοκράτες να τους ε, ε, απειλούμε ότι θα σας δίδουμε μόνο. Πρέπει να κάνουμε και δράσεις. Κυρία, κυρία έτσι. Όσον αφορά αυτές τις απάνθρωνες μεταχειρήσεις σε καμία περίπτωση μπορούμε να τις δεχτούμε σαν μέθοδο καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα πρέπει να στείλουμε λοιπόν ένα σαφές μήνυμα. Καταδικάζουμε κάθε είδους τέτοια επιχείρηση, είτε πρόκειται για τις δικές μας υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, είτε πρόκειται για αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και αν θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικές πρακτικές Γνωρίζω ότι κάποιοι από τους πολίτες των χωρών μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν επιθέσεις τρομοκρατικές είτε εικόνες από αυτές τις ε, φρικαλές ε, τρομοκρατικές επιθέσεις ότι μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι δυνατόν να δεχτούμε τέτοιου είδους πρακτικές. Πρέπει να τις καταδικάσουμε και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τις δεχθούμε. Είναι αντίθετες με τις αξίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, θα δώσω το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και προηγουμένως, πρόκειται εδώ για θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τα θέματα αυτά και θα ήθελα να ενθαρρύνει τα κρατημέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε ποτέ να μην προκύψει μια τέτοια υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κέντερς. Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων συμφωνήσαμε όλοι, χωρίς εξαίρεση, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση του τρόμου είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει δικαίωμα για την οποιαδήποτε παραπίαση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συνεχίζουμε να καταπολεμούμε και την τρομοκρατία σήμερα και να αντιμετωπίζουμε αυτές τις επιθέσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικές οι δηλώσεις που έγιναν σήμερα εδώ για να ξαναθυμηθούμε τι έγινε. Η άποψη του Συμβουλίου, πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή την πολιτική του Προέδρου Ομπάμα για να βελτιώσει την κατάσταση και όσον αφορά τα βασανιστήρια και όλες αυτές τις παράνομες ε, τεχνικές ανακρίσεων. Βεβαίως ε, σας άκουσα πολύ προσεκτικά κυρία Ίνφελτ και όλους όσους θέλουν να επικρίνουν με αυστηρότητα το Συμβούλιο. Όμως το Συμβούλιο δεν είναι υπεύθυνο για αυτά που συνέβησαν. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξουν ανακρίσεις, να υπάρξουν έρευνες, να αποκαλυφθεί η αλήθεια για το τι έγινε. Όμως δεν είναι αλήθεια ότι παρεμποδίστηκαν αυτές οι έρευνες, δεν υπήρξαν ε, δηλώσεις. Η μόνη δήλωση που έγινε ήταν μετά την 11η Σεπτεμβρίου όταν το Συμβούλιο δήλωσε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θέλω να μου βρείτε ποιες είναι οι δηλώσεις στις οποίες αναφερθήκατε που προέρχονται από το Συμβούλιο και που ε, δικαιολογούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεργασία σε αυτό το τομέα. Βεβαίως και πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά που είπατε ότι πρέπει ε, να βρεθούν ε, οι υπεύθυνοι και ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξει εδώ έρευνα και αλήθεια. Όμως είναι άδικο να κατηγορείται το Συμβούλιο και πολύ θα ήθελα εγώ να φτάναμε σε ένα άλλο συμπέρασμα ότι βεβαίως υπόλογοι υπάρχουν, ότι θα πρέπει να βρεθεί η αλήθεια, ότι σε κάθε περίπτωση στην Ευρώπη έχουμε ένα πολύ ισχυρό νομοθετικό και νομικό σύστημα και ότι αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γίνουν δεκτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι εμείς θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στηρίζουμε και τις αποφάσεις, τις πρόσφατες αποφάσεις του Προέδρου Ομπάμα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν εδώ δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να κατονομάζουμε υπεύθυνου οι οποίοι δεν είναι υπεύθυνοι, αλλά να ψάξουμε και να βρούμε τους πραγματικούς υπεύθυνου και την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. τέλος της συζήτησης.